τους υγειονομικού όρου που εφαρμόζονται στου μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσει ζώνης συντροφιά. Για να αρχίσουμε τη ζήτη, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Τέσσερα λεπτά. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, ο κασμός αυτός ε, τροποποιεί την ε, νομοθεσία που υπήρχε ήδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις για ηγέτρες κ. Φασούλη, Βίλιαμς, Παλέ, Νίκολσον, Εύεν και Ρόσπαχ για την εργασία τους ε, κατά τη διάρκεια των πολυπλοκών διαπραγματεύσεων. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και τις υπηρεσίες συναπόφασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Επί της ουσίας υπάρχει συμφωνία στην Επιτροπή Περιβαλλοντος αρχές Δεκεμβρίου και από τις αρχές του έτους ε, εξετάζουμε την εφαρμογή του άρθρου 290 για το θέμα αυτό. Καμιά φορά είχαμε την εντύπωση ότι δεν θα πετυχαίναμε να συμφωνήσουμε τελικά, το πετύχαμε όμως. Πετύχαμε μια συμφωνία και εξασφαλίσαμε έτσι ε, οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να μπορούν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα με τα ζωάκια τους και προβλέψαμε ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα ούτω ώστε ορισμένου χώρε να μπορούν να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα για 18 μήνες ανάλογα με την ασθένεια. Η οδηγία αυτή εξασφαλίζει οι βελτιώσεις να πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη. Παρατείνει το μεταβατικό καθεκτός μέχρι την 21η Δεκεμβρίου του 2011 για πέντε χώρες μέλη και από την 1η Ιανουαρίου του 2012 θα αναγνωστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπεται επίσης ε, το μεταβατικό καθεστώς να συμπεριλαμβάνει την εχινοκοκίαση και τα τσιμπούρια και να έχει την ίδια παράταση μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2011. Όσον αφορά τη διαδικασία της επιτροπολογίας, θα πρέπει η Κομισιόν να μπορεί να αναλάβει για τους στόχους αυτού του κανονισμού να βασιστεί στο άρθρο 290 το Συμβούλιο θα μπορούσε να μεταβάσει στην ε, ε, Κομισιόν τη δυνατότητα υιοθέτησης μη νομοθετικών πράξεων για την ε, οδηγία αυτή. Παραδείγματο χάρη για τον έλεγχο άλλων ασθενών εκτός από τη λίστα. Η Κομισιόν θα μπορεί να εφαρμόζει τα άρθρα που που ε, ε, παίζουν εδώ ένα σημαντικό ρόλο να μπορεί να τρομοδοποιηθεί η οδηγία αν υπάρχουν τεχνολογικές εξελίσεις και επίσης να τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές για το αντιληστικό εμβολιασμό για να ληφθούν υπόψη πρόοδος τεχνολογική και επιστημονική που ενδεχομένως θα επιδεχθεί μέχρι τότε. Συμφωνήσαμε στη διατύπωση για την εφαρμογή του άρθρου 290 και αυτό είναι σύμφωνο με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στα πλαίσια της Εθήκης Λισαβόνας. Η συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση κατέδειξε πόσο κατεπήγον είναι το θέμα. Θα ήθελα να πω ότι δημοκρατικά έχουμε εδώ δώσει ένα σημαντικό μήνυμα που θα πρέπει να μας κάνει να είμαστε περήφανος σαν σώμα γιατί η συγητή από μια μικρή πολιτική ομάδα μπόρεσε να έχει τόσο σημαντικό θέμα και να έχει τη συνεργασία των ισχυωδών εισηγητών από άλλε ομάδε. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να σα ευχαριστήσω όλου και επίση του εκπροσώπου από την Κομισιόν, το ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό και ελπίζω οι συνάδελφοι να μα υποστηρίξουν. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο ε, Επίτροπο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για το θέμα αυτό και ιδιαίτερα την εισηγήτρια την κυρία Ντεμπρούν για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να φτάσουμε σε συμφωνία ε, επί του θέματος το οποίο είναι αρκετά λεπτό για ορισμένα κράτη-μέλη. Πέρα από τα εμπλεκόμενα ζητήματα, έπρεπε να εκκινήσει μία διαδικασία σε σχέση με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης και την ευχαριστώ γι' αυτό. Οι εντατικές συζητήσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων οδήγησαν σε ένα κείμενο συμβιβασμού το οποίο αντικατοπτρίζει τα τεχνικά μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τις ε, προσαρμογές που επιβάλλονται δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό κατά τρόπο αποδεκτό. Η κοινή μας εργασία ήταν περίπλοκη και επιβραδύνθηκε από αυτή την ευθυγράμμιση. Όμως το Συμβούλιο ε, όρισε αυτή την εργασία γέρος. Ως προς το, το κείμενο συμβιβασμού θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή δεν θα προτείνει περαιτέρω παράταση της μεταβατικής περίοδου που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2011. Αυτό σημαίνει ότι θα ισχύσουν εναρμονισμένοι κανόνες από την 1η Ιανουαρίου 2012. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού πριν από την 30η Ιουνίου 2011 ως προς την ανακοίνωση των κατεξουσιοδότηση πράξεων θα λάβουμε υπόψη όλα τα δεδομένα έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβουλίο να μπορέσουν να ασκήσουν τις εξουσίες όπως ορίζει το χρονοδιάγραμμα. Τέλος, η Επιτροπή δέχεται την κοινή της δέσμευση έτσι ώστε να μην προδικάσουμε την περαιτέρω διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης σε σχέση με μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις που ενέχουν τέτοιες διατάξεις. Ελπίζω να δεχτείτε το κείμενο συμβιβασμού το οποίο αντικατοπτρίζεται σε όλες τις ανησυχίες. Ευχαριστούμε κύριε Ντάλη. Τώρα έχουμε ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων Φιέλνερ, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση αυτή εν μέρη διότι προσπαθεί να διευκολύνει τη μετακίνηση ζώων συντροφιάς. Ταυτόχρονα προσπαθεί να εξασφαλίσει η νόση των ζώων να μην καλύψουν όλη την Ευρώπη. Όντας Σουηδός πρέπει να σας πω ότι ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ για αυτό το θέμα διότι έχουμε δύο ασθένειες που δεν έχουμε ευτυχώ στη Σουηδία. Η μία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι η λύσα. Δεν υπάρχει στη χώρα μας. Ε, καθώς προχωρούσε λοιπόν η εξέταση αυτής της έκθεσης, μας ανησύχησε ότι ε, μπορεί να έχουμε προβλήματα στη Σουηδία με αυτή τη ρύθμιση, δηλαδή μπορεί να μεταδοθεί η νόσος αυτή. Στη Σουηδία ε, έχουν δικαίωμα οι πολίτες να κάνουν κάμπινγκ όπου θέλουν. Ε, ευχαρίστως Βεβαίως ε, έχουμε και εξαιρέσεις για να μην έρθουν αυτές οι ασθένειες στη Σουηδία. Υπήρχε κάτι αρκετά προφανές στη συζήτηση. Η διαδικασία της επιτροπολογίας μπορούσε να δημιουργήσει κενά. Και αυτά τα κενά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μετάδοση αυτή τη νόσου τη ΒΙΔΙΑ. Ευχαριστώ λοιπόν όλου αυτού που εργάστηκαν πολύ σκληρά εφευρίσκοντα λύσει, διευκολύνοντα τη μετακίνηση των ζώων συντροφιά, αλλά διατηρώντα τι παρεκκλήσει που έχουν νομοθετήσει ορισμένε χώρε για να προστατεύσουν τι χώρε του. Δεν θέλουμε δηλαδή νέε ασθένειε να φτάνουν σε χώρε που είναι ελεύθερε από αυτέ τι νόσους. Ο κύριος Μακάβαν για τους σοσιαλιστές και Δημοκρατία. Η κυρία, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Ντεμπούν για αυτό για αυτή την έκθεση. Πιστεύαμε αρχικά ότι ήταν ε, απλός αυτός ο φάκελος, αλλά τελικά οδηγηθήκαμε σε μεγάλες διαπραγματεύσεις. Τη συγχαίρω λοιπόν και συγχαίρω και την Κομισιόν και τον Επίτροπο που ε, βρήκαν λύση συζητήσαμε σε βάθος τις τεχνικές πτυχές αυτής της νομοθεσίας. Αλλά η νομοθεσία αυτή έχει μεγάλη σημασία για πολλούς πολίτες και την ελεύθερη κυκλοφορία τους με τα ζώα συντροφιάς. Όταν αρχικά είχαμε υιοθετήσει α, ρυθμίσεις πριν από μερικά χρόνια, ε, ε, υπήρξε μια ευνοϊκή τάση, αλλά είχαμε και παρεκκλήσεις για την προστασία των χωρών που ήταν ελεύθερες από αυτές τις νόσους. Όταν τελειώσει η μεταβατική περίοδος και θα έχουμε τη νέα νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη, θα έχουμε εξασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο υγείας ε, και ευημερίας των ζώων. Ως προς την επιτροπολογία, υποστηρίζουμε την, ε, τον συμβιβασμό που ε, διαπραγματεύτηκε. Ε, θέλουμε ισότητα μεταξύ ε, Κομισιών και Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου για την, ε, τα νομοθετικά θέματα. Όταν μιλάμε για εμπειρογνώμονες στους οποίους πρέπει να συμβουλευτούμε, θα πρέπει να αναφερόμαστε στους εμπειρογνώμονες από όλες τις πλευρές, δηλαδή τα κράτη-μέλη, ΜΚΟ και εμπειρογνώμονες που συστήνει και το Ευρωκοινοβούλιο. Όλοι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνονται. Χαίρομαι που έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τη μεταβατική περίοδο και περιμένουμε τις νέες προτάσεις της Κομισιόν για μελλοντικά νομοθετήματα. Η κυρία Βαλέαν τώρα για τους φιλελευθέρους και τους δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, ας μην ξεχνάμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία είναι θεμέλιο της αγοράς για την ενίσχυση του ανταγωνισμού της οικονομίας ευρείας κλίμακας και την προσέλκυση κεφαλαίων. Εν τω μεταξύ η ελευθερία της κυκλοφορίας για τους ανθρώπους είναι βασικό συστατικό μέρος και θεμελιώδες δικαίωμα. Έχουν καταργηθεί πολλά εμπόδια εθνικά και οι Ευρωπαίοι πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποφεληθούν. Έτσι οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν και τα ζώα συντροφιάς χωρίς να υπάγονται σε ιδιαίτερους κανόνες. Αλλιώς δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν. Χαίρομαι που ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση η Κομισιόν. Χαίρομαι για το γενικό καθεστώς διαβατηρίου που εναρμονίζει τις συνθήκες και τους όρους και βοηθάει την κινητικότητα των ζώων συντροφιάς. Συμφωνώ όμως ταυτόχρονα ότι πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Αυτό το μεταβατικό καθεστώς θα μας δώσει τη δυνατότητα να θεσπίσουμε τη σωστή υποδομή. Οπωσδήποτε είμαι σίγουρη ότι θα, αύριο θα υπερψηφίσουμε την παράταση της μεταβατικής περίοδου σε ορισμένα κράτη-μέλη, καθώς αυτά τα κράτη-μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένους κινδύνους. Δεν είναι η πρώτη φορά που ορισμένες χώρες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυστηρότερα μέτρα. Αρχικά τον Ιούλιο του 2008 έπρεπε να λήξει η μεταβατική περίοδος, επεκτάθηκε για το 2010. Τώρα έχουμε νέα επιμήκυνση. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες των κρατών που θεωρούν ότι η νόση είναι ε, πρόβλημα για αυτές. Και χαίρομαι που θα γίνουν και προγράμματα εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξάλληψη της λύσας. Φαντάζομαι ότι αυτή πρέπει να είναι η τελευταία ε, παράταση της ειδική μεταχείρισης ορισμένων χωρών. Ασυμμετρικά μέτρα θα φέρουν τα ωφελήματα που θέλουμε. Η, η μεταβατική περίοδος θα πρέπει να περιοριστεί συνεπώς και να έχουμε ισότητα σύντομα. Το πιο αμφισβητούμενο θέμα στην έκθεση δεν είναι το περιεχόμενο. Προκλήθηκε έντονη συζήτηση για την εφαρμογή των, ε, της συνθήκης της Λισαβόνας ε, για την επιτροπολογία. Είναι η πρώτη συναπόφαση, αν θέλετε, που πρέπει να εφαρμόσουμε τους νέους όρους. Αυτός ο κανονισμός δεν πρέπει λοιπόν να δημιουργήσει κακό προηγούμενο για μελλοντικέ αποφάσεις. Γι' αυτό η γραπτή συμφωνία κατά τον τρίλογο είναι σωστή ε, και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο αυτό το θέμα. Ο κύριος Νίκολσον για τους συντηρητικούς και τους μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον την εισηγητρία για όλη τη σκληρή δουλειά και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά υποστηρίζω αυτό που είπαν πολλοί από εμά, δηλαδή ότι αρχικά νομίζαμε ότι αυτό ο φάκελο θα ήταν απλός, χωρίς μεγάλα προβλήματα και τελικά ε, έγινε πολύ πιο επικίνδυνο ζήτημα ε, η συγγήτρια χρειάστηκε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις και να εργαστεί πολύ σκληρά για να περάσει η έκθεση μέσα στο σωστό χρονοδιάγραμμα επειδή υπήρχε πίεση για την επέκταση, την παράταση μιας παρέκκλησης που έλεγε τον Ιούλιο. Είναι ζωτικό νομοθέτημα αυτό λοιπόν, το οποίο θα βοηθήσει τα κράτη που ανησυχούν για τη λύσα. Η λύσα εξακολουθεί να εμφανίζεται σε ορισμένε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε ότι οι καμπάνιες εμβολιασμού θα βοηθήσουν στην εκρίζωση. Μέχρι τότε έχουμε βρει ένα τρόπο που μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τις προϋποθέσεις της μεταβατικής περίοδου χωρίς να ευθυγραμμίσουμε άμεσα ε, τη συμπεριφορά όλων των κρατών μελών. Η κυρία Ρόσμπαχ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νεμπλούν για την εργασία που επετέλεσε για το θέμα αυτό που ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ δύσκολο να ε, ταξιδέψει κανένα στην Ευρώπη με το κατοικίδιο ζώο του συντροφιάς. Ε, υπάρχει γραφειοκρατία τόσο πολύ που δυσκολεύει το ταξίδι, το κοινό ε, της, ε, μιας οικογένειας μαζί με το ζώο της. Βέβαια είναι δύσκολη η, γραφειοκρατία αλλά και απαραίτητη και γι' αυτό πολλές χώρες προσπαθούν να καταπολεμήσουν διάφορες αρρώστιες ε, των ζώων ε, ιδίως στην περίπτωση της λύσας καμιά φορά υπάρχουν προγράμματα υποχρεωτικής ε, καταναγκαστικής ε, εξαρτίας εμβολιασμού των άγριων ζώων και θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση με τα δικά μας. Η προστασία δεν σημαίνει καταστροφή και ελπίζω και άλλοι να μας μιμηθούν στις προσπάθειές μας και δεν ξέρω θα μπορούσε να μου πει η Κομισιόν να θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα να ξανεισαχθούν οι κτηνιατρικοί έλεγχοι στα σύνορα, ώστε ένα ιδιοκτήτη ε, κατοικιδίου ζώου να μπορεί να αποδείξει ότι εισαγάγει ένα ζώο το οποίο είναι εμβολιασμένο και είναι απόλυτα υγιές. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για χείρους, για άλλα ζώα ε, που δεν θα χρειάζεται να περνάνε απαρατήρητοι όπως αυτή τη στιγμή καμιά φορά γίνεται λάθρεμπόριο μικρών ε, σκύλων ή γατών. Ευχαριστώ Λεπρός. Δύο λεπτά κύριο Σνέλχαλτ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας χαιρετίζουμε και σας καλωσορίζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την εισηγήτρια, η οποία εργάστηκε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι το έγγραφο αυτό καλύπτει πάρα πολλούς τομείς. Βέβαια, τα περασμένα χρόνια είδαμε να υπάρχει αύξηση του αριθμού των κατοικιδιών ζώων και της επιθυμίας για τη μεταφορά τους πέρα από τα σύνορα. Είναι σωστό αυτό. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο για τον ιδιοκτήτη να μπορεί να πάρει το ζώο της συντροφιάς μαζί του. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να αποφύγουμε την διεύρυνση και την εξάπλωση ασθενειών στην Ευρώπη. Έχουμε καλές οδηγίες παραδείγματο χάρη 1998 του 2003 και από το 2012 θα υπάρχει το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ασθενειών που θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα ζώα αυτά εμβολιαστεί και επίσης ε, θα υπάρχει και ο ηλεκτρονικός έλεγχος από το 2011 και μετά. Κυρίε και κύριοι, πολλά κάναμε για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τις επιζωοτίες ε, στην Ευρώπη, ιδίως ε, όσον αφορά το θέμα της λύσας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε το θέμα του εμβολισμού των αλεπούδων. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Απ' την άλλη μεριά, οι εξτακτοί κανόνες που εγκρίνονται συνεχώς για κάποιες χώρες επιβαρύνουν τους πολίτες. Εγώ δεν βλέπω ότι υπάρχει ανάλογο όφελος με την επιβάρυνση. Πολλοί πολίτες μου έγραψαν με παράπονα για ε, πάρα πολύ δύσκολη συμπεριφορά στα σύνορα παράδειγμα Μεγάλη Βρετανία. Κάποιος πήγε να ε, ε, εισέλθει στη χώρα αυτή δύο μέρες πριν από αυτό που είχε δηλώσει. Το αποτέλεσμα ήταν μια, ένα πρόστιμο 3.000 ευρώ και κρατήθηκε το ζώο έξι εβδομάδες σε καραντίνα. Ε, αυτά είναι πολύ υπερβολικά πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να έχουμε κοινού κανόνες για όλους και να μην επιβαρύνουμε τους ιδιοκτήτες των κατοικιδίων αυτών ζώων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ο Γιολάινεν, δύο λεπτά επίσης. Μάλιστα. Ε, κύριε Επιτραπενταλή, σα καλωσορίζω στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον συναδελφό Σνέλχαρτ. Γι' αυτό έχετε πολύ μεγάλο έργο να αντιμετωπίσετε στο τομέα μέχρι το 2011. 11 θα πρέπει να δημιουργηθούν ίδιες προποθέσει και στι 27 χωρί μέλη ούτως ώστε τα ζώα συντροφιάς αυτά να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς πρόβλημα από τη μία χώρα στην άλλη. Ελεύθερη κυκλοφορία για τους σκύλους και τις γάτες ήταν ο στόχος της οδηγίας του 2003. Τώρα για τρίτη φορά προβλέπουμε μία εξαίρεση. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά ορισμένα πράγματα διαρκούν πάρα πολύ. Δέκα χρόνια για να προσαρμοστούν οι κανόνες αυτοί. Καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει την εισαγωγή ε, ασθενειών και γιατί 22 χώρες να το δέχονται να ταξιδεύει κανένας με τη γάτα ή το σκύλο του και 5 χώρες όχι Και εξετάστε το σας παρακαλώ για να δείτε κατά πόσον η πραγματικότητα είναι σύμφωνη με τις έκτακτες αυτές διατάξεις γιατί ξέρω ότι υπήρξαν πάρα πολλές ε, συζητήσεις, είμαστε όμως ένας χώρος δικαίου και το αργότερο το 2011 θα πρέπει να ε, πραγματοποιήσουμε την εσωτερική αγορά για τα κατοικίδια ζώα και τα ζώα της συντροφιάς. Ε, ε ο από κύριο Σνέλχατ ότι θα υπάρχει αυτό το διαβατήριο των εμβολιασμών και ο ηλεκτρονικός έλεγχος όταν κανένας ταξιδεύει με το ζώο του για διακοπές ή για να πάει στην εργασία του. Αυτός ο κανονισμός για τα κατοικίδια εδώ θα περάσει στην ιστορία γιατί είναι η πρώτη νομοθετική πράξη μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και θέλουμε να είμαστε επίσης όρις με το Συμβούλιο των Υπουργών όταν αναθέσουμε στην Κομισιόν το θέμα αυτό ήταν σκληρή ο αγώνας άξε κόπο. Ευχαριστούμε κύριε Αντιβρούν για την έκθεσή σας και για αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία. Να ξεκινήσει δηλαδή έτσι καλά έχουμε 100 νομοθετικής ε, πράξεις το χρόνο έχουμε 6.000 όμως μ, ανατεθειμένες θέσεις σας ευχαριστώ πολύ σας ευχαριστώ και εγώ ο κύριος Ντέιβις Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και Επίτροπε. Θα ήθελα να επικροτήσω την νομοθεσία που φτιάξαμε. Καταλαβαίνω ότι βασίζεται πάνω στις διατάξεις του Ηνωμένου Βασιλείου που εισήχθησαν πριν από 10 χρόνια. Η καραντίνα όμως στη χώρα μας έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και στα ζώα και στους ανθρώπους ο Φρόντο Μπάγκενς, ένας σκύλος ήταν ο πρώτος ο οποίος ταξίδεψε ελεύθερα και μετά χιλιάδες άλλα ζώα ακολούθησαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν εισήγαγε την ίδια νομοθεσία πριν από πέντε χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Εκατοντάδες χιλιάδων ζώα συντροφιάς ταξιδεύουν σήμερα στην Ευρώπη. 60% ε, είναι βρετανικά ζωάκια. Ε, αυτό κάτι λέει για το χαρακτήρα των Βρετανών, αλλά ας το αφήσουμε η ισορροπία είναι σωστή. Δηλαδή θέλουμε κινητικότητα χωρίς εξάπλωση των ασθενειών. Η λύσα είναι υπό έλεγχο. Έχουμε κατέβει σε λιγότερο από 300 περιπτώσεις πέρυσι και ούτε μία περίπτωση που να έχει να κάνει με την κυκλοφορία των ζώων. Λυπάμαι Ε, που η αριθμή κυκλοφορίας δεν είναι τόσο υψηλή όσο περίμενα. Πολλοί ιδιοκτήτε στην Βρετανία με ρωτούσαν αρχικά γιατί δεν ε, συμπεριλήφθησαν και άλλα ζώα για εκθέσεις όπως τα φέρετς ας πούμε μπορούν να εμβολιωστούν για τη λύση, αλλά δεν ε, καταδεικνύεται αυτό Τέλος πάντων, η λύση σε αυτά τα ζώα ήταν τόσο μικρή, ε, τόσο χαμηλή, ώστε μπορούσαμε να τα περιλάβουμε. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Πορτογαλία, τα ζώα αυτά, τα φέρετς, δημιουργούν κάποια θέματα και κύριε Επίτροπε για να τελειώσω θα ήθελα να πω ότι είναι οι φίτσε είναι αυτά τα ζώα, τόσο σωρό θα του ταλαιπωρώ με αυτό. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι σχόλιο τη Διερμηνέα. Λοιπόν, α, χαίρομαι που περιλήφθησαν και οι νηφίτσες, διότι έτσι μπορούν να κυκλοφορήσουν και τα σκυλιά και τα χατιά και οι νηφίτσες. Ο κύριος Βόιτσεκ είναι ο επόμενο ομιλητή. If he is not here, I will give floor to Mr. Agnew. δεν είναι εδώ, περνάμε στον κύριο Άγνιου. Κατανοώ ότι η αρχική ιδέα ήταν να έχουμε διαβατήρια ε, για τα ζώα συντροφιάς. Από το πιο τρελό κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου ε, προήλθε αυτό. Αρχικά υπήρχε περίοδος ε, καραντίνας έξι μηνών, αλλά με αυτό το νέο διαβατήριο δεν μπορεί να γίνει διάδοση, δεν υπάρχει πιθανότητα διάδοση των ασθενειών. Έτσι, η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούσε να προωθήσει την άρση της καραντίνας με αυτά τα διαβατήρια. Βεβαίως τα εμβόλια δεν σημαίνει ότι με την ύπαρξη εμβολίων δεν σημαίνει ότι δεν, δεν ε, διαδίδονται οι αρρώστιες διασυνοριακά γιατί πολλές φορές ε, μπορεί να γίνει εμβολιασμός ενός ζώου το οποίο είναι φορέας της ασθένειας χωρίς να φέρει τα συμπτώματα. Και πολλές φορές δεν υπάρχει τυποποίηση αυτού του προγράμματος. Άλλοι θέλουν επίσημο διαβατήριο, ενώ άλλα κράτη θέλουν οποιαδήποτε τεκμηρίωση. Άλλοι δεν δέχονται το διαβατήριο ως απόδειξη εμβολιασμού. Ορισμένες αερογραμμές αλλάζουν τη διαδικασία. Με άλλα λόγια, περιμένουμε να συμβεί ένα ε, ατύχημα πριν δράσουμε. Δυστυχώς αυτό έχω να πω και μόνο στην Επιτροπή. Ο κύριος Ντέιβις με την πλέ καρτέλα κάτι θέλει να πει. δεν νομίζει ότι ο φιλιππικός του θα ήταν καλύτερος ε, εάν είχε χρησιμοποιήσει αυτή, η χώρα του αυτή τη νομοθεσία πριν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλούς πολιτισμούς, είναι πολύ μεγάλη και δεν εμπιστεύουμε αυτό το σύστημα, λέει ο κύριος Άγνιου, και θα επιδεινωθεί η κατάσταση να το ξέρετε. Η ε, κυρία Μαγκίνες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Καλωσορίζω και τον Επίτροπο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Και όπως είπε ο κύριος Άγνιου, περιμένουμε να γίνει ένα τύχημα πριν δράσουμε. Τι κάνουμε δηλαδή, επεκτείνουμε τις, ε, ε, επεκτείνουμε τις εξαιρέσεις, αλλά αυτό που θα έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να υπάρχει διακίνηση των ζώων συντροφιάς λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες ε, προδιαγραφές υγείας και υγιεινή. Χρειάζονται λοιπόν αυστηροί έλεγχοι, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί θέλουν να μεταφέρουν τα ζώα σύντροφιά ε, όπου πηγαίνουν, όπως πολλοί Βρετανοί. Βέβαια, πώς θα έχει ζωή μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, αναρωτιόμαστε. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας και η συγγήτρια έθεσε το θέμα πολύ σωστά και τη συγχαρήκαμε γι' αυτό. Εάν όμως δεν προβλέπονταν μέτρα για να ανταποκριθείτε στις ανησυχίες της Ιρλανδίας, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, τι θα κάνατε. Το μέλλον είναι πολύ πιο σημαντικό. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι θα δείτε πώς εξελίσσεται η νέα νομοθεσία και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει σε αυτό το στάδιο. Θέλουμε οι υψηλές προδιαγραφές υγείας και υγιεινής για τα ζώα και τους ανθρώπους. Να συγχαρούμε λοιπόν την εισηγήτρια και όλους τους εμπλεκόμενους. Πιστεύω ότι ικανοποιήθηκαν οι περισσότερες ανησυχίες όχι βεβαίω τη αριστεράς πτέρυγα και ελπίζω να προβλέψετε μία νέα νομοθεσία για τη μεταφορά ζώων συντροφιάς. Υπάρχει νομοθεσία για ζώα αγροκτημάτων, αλλά όχι για ζώα συντροφιάς. Η κυρία Ούφσκοκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή έχει υποβάλει μια πολύ καλή πρόταση για να τροποποιηθεί ο κανονισμός ε, για τους κανόνες υγιεινής που διέπουν τη μεταφορά ζώων συντροφιάς. Ελπίζω να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος για αρκετές χώρες μεταξύ αυτών και η Σουηδία για να αντιμετωπιστεί το θέμα, η ασθένεια της λύσας που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέπονται ειδικοί έλεγχοι και οι ασθένειες όπως η εχινοκοκίαση θα μπορούσαν να επεκταθούν στη Σουηδία και αυτό θα ήταν επιζήμιο για την ελεύθερη μεταφορά για μια χώρα όπως η Σουηδία. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε διότι αυτή η προσωρινή λύση επετράπη μετά από προσπάθειες της συζήτητρες και άλλων. Η επόμενη ομιλήτρια για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, τη συνάδελφο Μπρουνιέ του σκληρή εργασία που έκανε για αυτή την εισήγηση. Πέθανε ε, ένας άνθρωπος πέρυσι από Λίσσα στην Ιρλανδία. Προσπαθούσε να σταματήσει ένα καυγά μεταξύ δύο σκυλιών στην Νότιο Αφρική και πέθανα από λύσα. Είχαμε και άλλη περίπτωση πρόσφατα και η λύσα είναι μία από τις πιο σοβαρές ασθένειες που επηρεάζει τους ανθρώπους. Ε, τα ταξίδια σήμερα σημαίνουν ότι η ασθένεια είναι πολύ κοντά στην πόρτα μας πάντοτε, γι' αυτό έχουμε αυστηρή καραντίνα και μόνο με αυτή την αυστηρή καραντίνα είμαστε ελεύθεροι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε. Γι' αυτό η μεταβατική περίοδος δεν θα πρέπει να τελειώσει το 2010 τον Ιούλιο. Οι διασφαλιστικές ε, ρήτρε είναι σημαντικές και για τα ζώα και για τους ανθρώπους. Πολεμούν τη λύσα αλλά και τα τσιμπούρια ε, τα οποία και αυτά δεν έχουμε στην Ιρλανδία. Δεχόμενη λοιπόν αυτή την πρόταση κύριε Πρόεδρε θα διευκολύνουμε τον αγώνα για την εξάλληψη της λύσας από την Ευρώπη. Είναι πήγον λοιπόν το ζήτημα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Και τώρα με τη διαδικασία Catch the Eye έχω τρεις ομιλητές. Ο κύριος Νικολάσετς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, συμφωνώ με ε, αυτό που ελέγχθη, δηλαδή όσον αφορά τις ε, κτηνιατρικές απαιτήσει που διευκολύνουν τη διέλευση των ε, ενδοκινοτικών σύνορων και καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν, της εισηγητρίας, της οποίας η εργασία είναι υψηλωτά του επίπεδου, όσον αφορά του συμβουλισμού κατά ε, της λύσας και άλλων ασθενειών και ελπίζω ότι αυτό θα συμβάλλει στην εναρμόνιση των κανονισμών για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο από ε, ασθένειες λύσας. Πολλοί από μας θέλουν να μεταφέρουν τα ζώα συντροφιάς τους και θα ήταν καλό νομίζω να παρατηθεί η εξαίρεση παραδείγματος χάνει για, για χώρες όπως η Ελλάδα που υπάρχουν πιο αυστηροί εσωτερικοί κανόνες. Θα πρέπει να έχουμε προληπτικά μέτρα και μου φαίνεται πάρα πολύ καλό αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Σαπιά, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της και να συγχαρώ ακόμη και όλους αυτούς που συνέβαλαν για το συμβιβασμό. Χαίρομαι που μπορούμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τα προστατευτικά μέτρα κατά της λύσας. Χαίρομαι ακόμη που θα έχουμε τη δυνατότητα όμως να επιτρέψουμε την κυκλοφορία των ζώων συντροφιάς μετά το 2011. Είναι καλό συμπιβασμός αυτός, δίνει αποτελεσματική απάντηση σε μια στιγμή όπου τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να ανησυχούν για ορισμένες ασθένειες ε, η Κομισιόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια εμπειρογνώμων από τα κράτη-μέλη, από ΜΚΟ και από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να προχωρήσει. Έχουμε γραπτή εγγύηση ότι δεν θα αποτελέσει η ρύθμιση αυτή προηγούμενο για το μέλλον. Έτσι, το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να ανησυχεί όσον αφορά τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας την ενδεχόμενη αξιολόγηση σαν προηγούμενο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μόλτσα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαλείψουν ε, τις επιζωοτήσει και τις ασθένειες του ζώνου στη Λίσσα είναι πάρα πολύ αξιόλογες και είναι πάρα πολύ θετικό να υπάρχουν κάποια μέτρα ούτως ώστε να μπορεί να είναι δυνατό ο τουρισμός με ε, Κάτι ζώα η ζώα συντροφιά. Νομίζω ο ηλεκτρονικό ε, έλεγχο, το ηλεκτρονικό διαβατήριο είναι κάτι πολύ θετικό. Από την άλλη μεριά, ξέρω από την Ευστρία ότι υπάρχουν ε, προβλήματα, παραδείγματο χάρη το λαθρεμπόριο ε, ζώων συντροφιά από φθηνέ χώρε της Ανατολική Ευρώπη ή από αλλού ε, και επίσης οι μαζικές μεταφορές ζώων ε, από τη μια άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη διαμετακομιζόμενες από την Αυστρία μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε ε, ασθένες. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε γιατί οδηγούν στη διεύρυνση επιζωτιών όπως στη Λίσσα. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο να έχουμε εδώ κάποια συγκεκριμένα μέτρα αποτρεπτικά. σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο να απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμοι βουλευτέ, ε, μπορούμε να είμαστε νομίζω όλοι περήφανοι για την γλίγορο πρόεδρο που ετεύχθη για το θέμα αυτό, που, πράγμα που έγινε υπό έντονη χρονική πίεση και σε δύσκολα νομοθετικά πλαίσια. Η παράταση κατά 18 μήνες ε, του καθεστώτος που, που διέπει τις μεταφορές των ζώων αυτών σε πέντε χώρες μέλη θα δώσει τη δυνατότητα προσαρμογής μέχρι τότε ε, για να μπορέσουν να υπάρχει εναρμόνιση με τις άλλες χώρες μέλη. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν προβλέπει περαιτέρω παράταση η Κομισιόν. Ταυτόχρονα η παράταση αυτή όμως θα επιτρέψει στην Κομισιόν να υποβάλει ε, μια συνολική πρόταση για την αναθεώρηση του συνόλου της οδηγίας και επίσης για την ευθυγράμμιση της παλιάς ε, διαδικασίας της επιτροπολογίας με την συνθήκη της Αβώνας. Συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τους πολίτες και χαίρομαι που ήταν ευτυχές στο τέλος. Πρώτα σε ευχαριστώ. Η κυρία Ντουμπρούν, η συγγήτρια να ολοκληρώσει. Μάλιστα, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ την παρουσία του Επιτρόπου Ντάλι στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο, να τον καλωσορίσω και να χαιρετήσω τη δυνατότητα συνεργασίας μαζί του. Ε, χαιρετήσω επίσης ε, την δήλωση που έκανε σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο όταν είπε ότι συμφωνήθηκε το περιεχόμενο με την Κομισιόν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω εκείνους που μίλησαν εδώ στην ε, συζήτηση, οι περισσότεροι υπέρ των συστάσεων, ορισμένοι κατά βέβαια. Θέλουμε να έχουμε μια προσέγγιση με επιστημονική βάση. Έχοντας κατά νου βέβαια την κατάσταση σε κάποια κράτη-μέλη όσον αφορά τους, ε, τη λύσα. Η Κομισιόν ε, έχει μια προσέγγιση προληπτική και ελπίζουμε ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν πόροι κοινοτικοί για να συνεχιστούν οι εκστρατείες εμβολιασμού κατά της λύσης σε ορισμένα κράτη-μέλη. Όπως είπε η Κομισιόν θα μπορούσε να αλλάξει η υποδομή, θα μπορέσουν να υπάρξουν ε, νέα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού που κάνουν τους αυτούς οι μεταβατικές ε, διατάξεις θα παραταθούν μέχρι τα τέλη του 2011 και μέχρι τότε οι διατάξεις για την διαμετακόμιση των ε, ζώων συντροφιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει εναρμονιστεί. Εν τω μεταξύ όλοι θα μπορούν να κινούνται στην Ευρώπη με τα ζώα τους. Βέβαια το μεταβατικό σύστημα θα επιτρέψει ορισμένα κρατημένα να έχουν πιο αυστηρά συστήματα από ό,τι άλλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με βοήθησαν σε αυτό το πολύ πολύπλοκο και δύσκολο έργο, αξιόλογο όμως σε τελευταία αναλύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you too, Ms. Ευχαριστώ την κυρία Ντεμπρόν και όσους συναδέλφους μίλησα. Έληξε η συζήτηση ή ψηφίζουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι για αυτό το θέμα. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Κομισιόν για